Hello everyone. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Καθίστε σας παρακαλώ πολύ για να ξεκινήσουμε και τη συνεδρίασή μας. Καταρχάς, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς κάποια τροποποίηση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Αρμόδιο για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια Υποθέσει και την Αλία, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Καλώ ήρθατε λοιπόν, Επίτροπε Βέλλα, στη συνεδρίασή μα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μα ενδιαφέρουν και επί των οποίων είστε εσεί αρμόδιο. Πραγματικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι γίνεται με την εφαρμογή του εβδόμου προγράμματο προγράμματος για το περιβάλλον, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, τι γίνεται με την ε, μόλυνση των υδάτων από φαρμακευτικές ουσίες. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μαζί σας προκειμένου να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα ζητήματα αυτά. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για την παρουσίασή σας. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ Αντίνα. Αξιότιμοι βουλευτές, καλό σας απόγευμα. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε για το διαφρομένο διάλογο ήταν 9η Μαρτίου. Έκτοτε πολλή δουλειά έχει γίνει από κοινού για την ολοκλήρωση νομοθεσία ό,τι αφορά τον Ιτράργυρο, τα ροχ και το πακέτο για τα απόβλητα. Ναι, θα δοθεί το πράσινο φως σε αυτή την οδηγία από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο. Οι κανόνες αυτοί για τα απόβλητα ενισχύουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πρωτοπόρο στο θέμα της διαχείρισης ε, και ανακύκλωσης αποβλήτων. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της πολύ καλής μας συνεργασίας. Σήμερα θα ήθελα να δούμε την ευρύτερη εικόνα όταν πρώτο ήρθα εδώ πριν από 3,5 χρόνια, τρεις προτεραιότητες όρισα. Πρώτη είναι η συνεισφορά μας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη. δεύτερη προτεραιότητα ήταν να έρθουμε εκ νέου σε επαφή με τους πολίτες και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Και τρίτη προτεραιότητα ήταν με την καλύτερη υλοποίηση να πετύχουμε αυτά αποτελέσματα στους τομείς αυτούς. Ε, και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι η Κομισιόν με τη δική σας βοήθεια έχει αποτελέσματα και στους τρεις ε, τομείς. Ε, έτσι το περιβάλλον της, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης ε, έχει βελτιωθεί και θα έχει βελτιωθεί όταν ολοκληρωθεί αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος. Πρώτη προτεραιότητα, ευθυγραμμισμένη και με τις προτεραιότητες της Κομισιόν συνολικά, ήταν πράσινη και γαλάζια οικονομία. Η πιο κυκλική οικονομία μεταξύ άλλων. Έχουμε πετύχει πολλά εδώ. Υπάρχει ευρεία συνένεση ως προς το σχέδιο δράση για τη κυκλική οικονομία του 2015, το οποίο πλέον εξορθολογεί και περιλαμβάνει σε όλες τις διαστάσεις της πολιτικής ε, τη διάσταση της κυκλικής οικονομίας. Ε, και στις ε, συζητήσεις και στη χάραξη πολιτικής, το 80% δε των 54 δράσεων, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Και το Γενάρη ολοκληρώθηκε μια δύο μέτρων που είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα στη μεταβατική αυτή διαδικασία. Δεν θέλω να αναλάβω αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος Κατάινα το Φεβρουάριο. Θα υπενθυμίσω απλά ότι η στρατηγική για τα πλαστικά αποτελεί ένα νέο όραμα για μια ε, φυή καινοτόμο βιώσιμη βιομηχανία πλαστικών όπου η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση θα ενσωματώνεται πλήρω ε, στο σχεδιασμό και την παραγωγή. Υπάρχουν πολλές σημαντικές ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη για αυτούς που ανακυκλώνουν στην Ευρώπη. τεράστιε δυνατότητες ώστε το πλαστικό τα απόβλητα από πλαστικό να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, νέα υλικά εδώ στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι το 2030 το αργότερο όλη η συσκευασία ε, που είναι από πλαστικό να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί. Έτσι θα βελτιώσουμε την ε, οικονομία αλλά και την ποιότητα της ανακύκλωσης των πλαστικών και αυτές τις ευκαιρίες θα τις ε, κάνουμε πράξη. Επίσης δημιουργούμε κάποια μέσα και εργαλεία για να προωθήσουμε τις επενδύσεις και την καινοτομία ώστε να κλείσει αυτό το χάσμα γνώσης και να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για την ανακύκλωση. Όλα αυτά πολύ θετικά βέβαια για την ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι τα πλαστικά μίας χρήσης είναι μία μείζον πηγή διαρροής πλαστικών στο περιβάλλον. 50% των ε, απορριμμάτων ε, στις ε, παραλίες μας ε, το θέμα αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο. Εξού λοιπόν και εργαζόμαστε σκληρά. Υπάρχει πρόταση για τα πλαστικά μια χρήση αλλά και για τα λευτικά εργαλεία. Θα είναι έτοιμη το Μάιο η πρόταση αυτή. Επίση, το πλαίσιο παρακολούθηση και το έργο σε ό,τι αφορά την επαφή μεταξύ χημικών προϊόντων ε, και αποβλήτων, οι τρεις αυτές ε, νομοθετικές πράξεις, ε, θέλουμε να συνδυαστούν μεταξύ τους για να μην χάσουμε την όθηση και την ορμή που έχει ε, η πρόσεχη κυκλικής οικονομίας. Οι προσεγγίσει κυκλική οικονομία αναγνωρίζονται και εκτό Ένωση, όλο και περισσότερο. Χρειάζεται μια παγκόσμια μετάβαση στο μοντέλο τη κυκλική οικονομία, σημαντικό ρόλο τη Ένωση για τη μετάβαση τρίτες των τρίτων χωρών. Αυτή η παγκόσμια μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα βοηθήσει και στην υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Αργότερα φέτο, στο πλαίσιο του διάσκεψη κορυφή ε, τη ομάδα των 7, θα συζητηθεί το πόσο το μέσο των πλαστικών θα μπορούσε να γίνει πιο κυκλικό και να μην μολύνουν του ωκεανού ε, τα πλαστικά. σω ένα χάρτη για τα πλαστικά στο πλαίσιο του G7 ε, θα συνεισέφερε στην καλύτερη παραγωγή, κατανάλωση και διάθεση των πλαστικών, όπω προβλέπει ο 12ο στόχο βιώσιμη ανάπτυξη και στρατηγική τη Ένωση για τα πλαστικά. Και τα δύο στηρίζουν την υλοποίηση του 14ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για τους ωκεανούς και χαίρομαι που για πρώτη φορά και οι ωκεανοί έχουν προεξάρχουσα θέση στο θεματολόγιο της ομάδας των 7. Αυτό θα βοηθήσει και σε συνέχεια της ε, πολύ επιτυχημένης ε, διάσκεψης που οργανώσαμε για τους ωκεανούς τον Οκτώβριο του 2017 που μας έδωσε και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να ηγούμεθα σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα περί των ωκεανών. Ήμουν χθες ε, στις βελγικές ακτές. Καθαρίσαμε τις ακτές με εκατοντάδες ε, προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ειδών που ε, περισυλλέξαμε κυριαρχούσαν τα πλαστικά μιας χρήσης ε, και, ε, και τα απόβλητα λευτικών εργαλείων. Αυτό δείχνει πόσο δουλειά χρειάζεται να γίνει ακόμη για να προστατεύσουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Πέρυσι είχαμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα για τους ωκεανούς. Για τον 14ο στόχο είχαμε την, ένωση, την διάσκεψη του ΟΗΕ τον Ιούνιο και έπειτα στη Μάλτα είχαμε εμείς οργανώσει τον Οκτώβριο ως Ένωση την διάσκεψη για τους ωκεανούς με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, σχεδόν 450 δεσμεύσεις με τρίσιμες τέσσερα. Πάνω από 7 δις ευρώ για δέσμευση υπόρων και 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, είναι οι πρόσθετες ε, θαλάσσιες πρωτευόμενες περιοχές. Η δεύτερη προτεραιότητα για μένα αυτής εξ αρχής ήταν να ε, αναλαμβάνω η προσέγγιση των πολιτών με την Ευρώπη, βελτίωση της ποιότητας των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν έχω δώσει πολύ μεγάλη σημασία στη βελτίωση της ατμόσφαιρας, του αέρα. <coughs> Ξέρουμε όλοι τι κινδύνους ενέχει η κακή ποιότητα του αέρα για την ανθρώπινη υγεία, η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τις ε, τιμές, τις ανώτατες τιμές στις εθνικές εκπομπές 2016, καθώς και άλλες σχετικές με την ποιότητα του αέρα ε, νομοθετικές πράξεις, όπως ε, η οδηγία για τα εργοστάσια καύσης, medium combustion plants, θα κάνει τεράστια διαφορά. Μέχρι το 2030 θα έχουμε μειώσει κατά το ίμιση τι αρνητικέ επιπτώσεις, αλλά είναι αργά το 2030 για τις 300.000 ανθρώπους που πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρώπη κάθε χρόνο λόγω κακής ποιότητα του αέρα ή για τα εκατομμύρια που υποφέρουν από άσθημα και άλλες ε, αναπνευστικές παθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν αναβαθμίσαμε τη δράση μα και ζητούμε από τα κράτη-μέλη ήδη από τώρα να ε, φροντίσουν ο να είναι πιο καθαρός και όχι σε 10 χρόνια. Έχουμε τους διαλόγους για το καθαρό αέρα που βεθούν τα κράτη-μέλη να μάθουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με μέτρα δοκιμασμένα αποδεδειγμένα, που αποδεδειγμένα λειτουργούν. Χρειάζονται βέβαια περισσότερες προσπάθειες. Πολλοί είναι ε, Πολλές είναι περιοχές στην Ευρώπη που ε, βλέπουμε απαράδεκτες ε, υπερβάσεις των προτύπων σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα αν δεν λάβουν ε, τα απαραίτητα μέτρα τα κράτη-μέλη για να μειώσουν στο δυνατόν αυτές τις υπερβάσεις ε, και χρονικά, πρέπει εμεί να αναλάβουμε δράση. Αυτό είναι ο ρόλο των διαδικασιών επί παραβάση. Και ήταν πολύ ξεκάθαρη και η Κομισιόν προ αυτό. Όταν τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα που περνάνε αποτελεσματικά έγκαιρα δεν έχουν ληφθεί, μετά και την επιλογική διάσκεψη που οργάνωσε για την ποιότητα του αίρεση 30 Ιανουαρίου, εμεί θα προχωρήσουμε και θα παραπέμψουμε τα εν λόγω κράτη-μέλη στο δικαστήριο. Τώρα που ολοκληρώθηκε η ενδελεχή ανάλυση όλων των συνεισφορών, μέσα Μαρτίου είχαμε υποσχεθεί και τήρησαμε το χρονοδιάγραμμα. Μπορώ να σα πω λοιπόν ότι θα προτείνω στο Σώμα των Επιτρόπων πράγματι να προχωρήσουμε μια σειρά ε, τέτοιων διαδικασιών επί παραβάση στο πλαίσιο του προσεχούς κύκλου διαδικασιών ε, επί παραβάση στα τέλη Απριλίου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου Στι διάφορε υπηρεσίε που εργάστηκαν σκληρά Του τελευταίους μήνες για την αξιολόγηση των στοιχείων. Ναι, είναι αξιοθαύμαστη η αφοσίωσή τους ανάγκες των πολιτών. Νερό τώρα. Και η προστασία αυτού του πόρου είναι πολύ ψηλά στο θεματολογιό μα. Το Γενάρη εγκρέαμε την πρόταση για το πόσιμο νερό. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα, θα προστατεύσει του καταναλωτέ από δυνητικέ μελλοντικέ απειλέ για την υγεία του και θα βελτιώσει την πρόσβαση στο νερό για όλου πρόταση περιλαμβάνει μια διάταξη για τη χορήγηση πρόσβασης ε, σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο πόσιμο νερό και έτσι ολοκληρώνεται η ανταπόκριση της Κομισιόν στην πρώτη επιτυχημένη ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών Right to Water, το δικαίωμα στο νερό παναχρησιμοποίηση του νερού είναι ένα άλλο πολύ ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση της σπάνιδος του νερού και εμείς ε, προσπαθούμε να αναπτύξουμε διάφορες δράσεις για να προωθήσουμε ε, μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα εστιάσουμε στην, ε, στον υπερκαρισμό των βασικών εμποδίων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπου αυτό βέβαια είναι αποδοτικός προς το κόστος και ασφαλές. Θα έχουμε μια νομοθετική πρόταση σύντομα για την άρδευση, τη χρήση δηλαδή του νερού ε, στη γεωργία. Θα την εγκρίνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ό,τι αφορά το REACH τώρα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ζωής έχει κάνει τη διαφορά τώρα την τελευταία δεκαετία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη σκέφτεται για τα χημικά. Δεν πρέπει αυτό να μα διαφεύγει. Πρόσφατα έγινε αξιολόγηση που αποδεικνύει ότι μετά από 10 χρόνια το REACH πλέον έχει βελτιώσει σημαντικά την προστασία τόσο τη ανθρώπινη υγεία όσο και του περιβάλλοντο. Επίση, έχει προωθήσει εναλλακτικέ ε, αντί, ε, αντί των δοκιμών ε, σε ζώα και έχει εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών στην ενιαία αγορά της Ένωσης. Το REACH λοιπόν πλήρωσε επιχειρησιακό και εκπληρώνει τους στόχους του. Βέβαια, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Ότι υπάρχουν κάποια κενά σε ό,τι αφορά τα δεδομένα ε, που θα πρέπει να καλυφθούν σε ό,τι αφορά του φακέλου καταχώρηση. Χρειάζεται ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών από την Ένωση και από τρίτε χώρε. Χρειάζεται μια πιο απλή διαδικασία αδειοδότηση, βελτιωμένη εφαρμογή τη νομοθεσία, περισσότερη στήριξη στο να μπορούν να συμμορφούνται στην νομοθεσία ΜΜΕ. Δεν μπορεί να τα κάνει όμω όλα αυτά η Κομισιόν. Στρέφομαι λοιπόν προς τα κράτη-μέλη και ζητώ μεγαλύτερη δέσμευση από πλευρά του, καθώ και τη διάθεση ενδεδειγμένων πόρων, ώστε πραγματικά να πετύχουμε τις βελτιώσεις αυτέ. Η φύση πάντοτε είναι ένα από του καλύτερου τρόπου διασύνδεση τη Ευρώπη με του πολίτε. Το Natura 2000 είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα τα προσθέμενη αξία. Χωρί τη φύση δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ποιότητα ζωή. Χαίρομαι λοιπόν που έχω να αναφέρω ότι η πρόοδο εδώ είναι θετική το σχέδιο δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία που εγκρίναμε πέρυσι τον Απρίλιο, πετυχαίνει και σε τις τέσσερις προτεραιότητες για την καθοδήγηση, το διάλογο και τη συμμόρφωση, τις επενδύσεις ε, και την ε, συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση. Θα έχουμε σύντομα νέα έγγραφα καθοδήγησης η ιδέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE για την διατήρηση φύσης στη βιοπικιλότητα αυξήθηκε κατά 10% και κάθε φορά που γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000, την 21η Μαΐου, βλέπουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να είμαστε όμως αυτάρες και όταν επαναπαυόμεθα. Το 2020 έφτασε. Πρέπει να κάνουμε πιο πολλά για να πετύχουμε τους στόχους σε ό,τι αφορά ε, τη βιοπικιλότητα. Μία μείζον πρόκληση είναι η ανησυχητική μείωση των επικονιαστών. Και γι' αυτό χρειάζεται επίγουσα ε, αποφασιστική δράση. Και σύντομα θα έχουμε καταθέσει τη σχετική πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα σε σχέση με αυτό που μας ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, πρωτοστατή και σε ό,τι αφορά την προστασία της ιοπικιλότητας, πέραν των εθνικών συνόρων. Μέσω των δεπατεύσεων BBNJ σε επίπεδο ε, ΟΗΕ. Το BBNJ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την παγκόσμια διακυβέρνηση των ωκεανών. Στόχο έχει την υλοποίηση και την ενίσχυση του, της UNCLOS, ώστε να τα αντιμετωπιστούν οι ειδικέ ανάγκες της συντήρηση, διατήρησης και βιώσιμη χρήση τη οπικιλότητας πέραν της εθνικής δικαιοδοσία. Τρίτη προτεραιότητα είναι πράγματι να τα πετύχουμε όλα αυτά που λέμε. Make it happen. Μόνο επιτόπου ε, βλέπουμε αυτά, αυτές τις πολιτικές και την νομοθεσία. Άρα πρέπει να εργαστούμε στην πράξη. Εξού και δουλεύουμε πολύ σκληρά ώστε όλοι αυτοί οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι στην πράξη. Ένα από τα νέα εργαλεία που αναπτύξαμε για αυτό το σκοπό είναι η περιβαλλοντική μελέτη υλοποίηση. Πέρυσι τη δρομολογήσαμε, καλύπτει μία διετία και ήδη επεξεργαζόμαστε τις εκθέσεις αναχώρα για το δεύτερο κύκλο 2019. Θα εγκριθούν σε 12 μήνες πρόθεσή μας είναι να προσθέσουμε τρία νέα θέματα. Την κλιματική αλλαγή, τα χημικά και τις ε, εκπομπές από τη βιομηχανία. Επίσης, ε, λαμβάνουμε περαιτέρω μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τη βασική, μία από τις βασικές αιτίες ε, της χαμηλής υλοποίηση που αναφέρεται στι εκθέσεις για την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι <clears throat> οι ανεπαρκείς μηχανισμοί αξιολόγηση της Συμμόρφωση και διακυβέρνηση. Το σχέδιο δράση, το σχετικό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη με τι πρακτικέ πτυχέ εξασφάλιση τη συμμόρφωση με καθοδήγηση παραδείγματο χάρη πάνω σε στρατηγικέ για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματο. Για όλα αυτά χρειάζονται σημαντικοί πόροι. Μεταξύ αυτών, βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, και χρηματοοικονομικοί πόροι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των συζητήσεων που συνεχίζονται για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο το επόμενο. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ακόμα τομέα που μπορούμε να συνεργαστούμε στενά για να ασκήσουμε χρήσιμη πίεση. Η μεταμόρφωση, αν θέλετε, του χρηματοοικονομικού πλαισίου είναι ένα εγχείρημα μεγάλη εμβέλεια. και ζητώ και χρειάζομαι την υποστήριξή σα ώστε να μπορέσουμε το κεφάλαιο να το ανακατευθύνουμε σε βιώσιμε δραστηριότητε. Εγκρίναμε στι 7 Μαρτίου ένα σχέδιο δράση για τα βιώσιμα οικονομικά που προβλέπει και έναν κανονισμό για ένα σύστημα ταξινόμησης ε, για ε, βιώσιμα οικονομικά. Στόχος μας, μάλλον μία δυνατότητα, είναι να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο του οικολογικού σήματος, το Eco Label, για ένα πρόγραμμα ετικετοθεσίας για κάποια χρηματοοικονομικά προϊόντα, ώστε οι επενδύσεις να γίνονται σύμφωνα με περιβαλλοντικές και κοινωνικές Παράμετρο και φυσικά θα σας στηρίσω ενήμερος για την πρόοδο στο θέμα αυτό. Έρχομαι στα μελλοντικά ε, κονδύλια. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο σχεδιασμός της τελικής αρχιτεκτονικής, αλλά εξετάζουμε το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σημερινή προσέγγιση, αλλά να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι σε όλα τα ταμεία, τα βασικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεσή σα για το 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντική δράση, επισημάνατε και πολύ σωστά ελλείψει στις πρακτικέ που ισχύουν σήμερα και συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτική πρέπει να είναι πιο, πιο συνεκτική και οι στόχοι, οι περιβαλλοντικοί θα πρέπει να ενταχθούν πιο επιτυχημένα στι υπόλοιπε πολιτικέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική που πρέπει να κάνει πιο πολλά για το νερό, τη φύση και τη βιοπικιλότητα ως έχει ε, στη σημερινή της μορφή δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Παρά το ότι έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση για τον οικολογικό προσανατολισμό και αυτό το επιβεβαιώνει και το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο. Γι' αυτό και λοιπόν απευθύνω έκκληση να διορθωθούν οι ανεπάρκειες στο πλαίσιο και των προσεχών μας προτάσεων. Η Κομισιόν επίσης προετοιμάσει και μια πρόταση για το πρόγραμμα LIFE μετά το 2020. Θέλουμε να ενισχυθεί ο ρόλος του σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ολοκλήρωση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα οποία εκμεταλλεύονται την ε, μόχλευση των κεφαλαίων από την κοινωνική πολιτική και την περιφερειακή πολιτική και προωθούν σχέδια και προγράμματα για το νερό, τον αέρα, τα απόβλητα και τη φύση. Χαιρετίζω την ε, μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα. Το έβδομο πρόγραμμα για το περιβάλλον ε, έχει έναν πάρα πολύ χρήσιμο σκοπό να υπηρετήσει. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε το πρόγραμμα συνολικά και προβλέπω, μάλλον έχω προγραμματίσει να γίνει μια ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς Περιμένω και τη δική σας υποστήριξη και προσβλέπω στην έγκριση αυτής ε, της ε, πρότασης στην Ολομέλεια. Βασίζομαι πάντα στη δική σας υποστήριξη ώστε η Επιτροπή σας να εξετάσει γρήγορα όλες τις νομοθετικές προτάσεις που παρουσιάσαμε θα παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες ώστε να ολοκληρωθούν ιδανικά πριν λήξει η θητεία αυτή του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ξέρω ότι μακρηγόρησα λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθω, αλλά ήθελα να σα δώσω μια πλήρη επισκόπηση ε, των τελευταίων 12 μηνών και τη πολύ σημαντική δουλειά που κάναμε. Φυσικά δεν μπορούσα να αναφέρω όλα όσα κάναμε και θα κάναμε του επόμενου μήνε. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα θέματα που παρήψα δεν είναι εξίσου σημαντικά και βεβαίω με ενδιαφέρει να ακούσω και τι δικέ σα προτεραιότητε. Σα ευχαριστώ λοιπόν και σα ευχαριστώ και για τη συνεχιζόμενη καλή σχέση που έχουμε όλη αυτή την περίοδο καθώς και την ε, επικοδομητική ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε. Ας ε, ακούσουμε τώρα τις ερωτήσεις καταρχάς από τους συντονιστές. Δύο λεπτά ο καθένας. Λίζε πρώτος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ποιότητα του αέρα. Μιλήσατε. Έχω μια ερώτηση. όλο και περισσότερο συζητείται αυτό το ε, νούμερο που επίσης μας αναφέρατε και εσείς για τους 400.000 πρόωρους θανάτους λόγω της ε, <clears throat> κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι, αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις μελέτες ε, που μιλούν για την ατμοσφαιρική μόλυνση δεν ξέρω κατά πόσον ε, είναι όμως ρεαλιστικό αυτό το νούμερο ε, των 400.000. Ξέρω ότι έχετε κινήσει διαδικασίες κατά διαφόρων κρατών μελών. Αν υπάρξει ε, προσφυγή ή αν υπάρχει καταγγελία, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει σε πέρα στα δικά της καθήκοντα και εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Σε κυρία Μπιακόφσκα, εγώ και κάποιοι άλλοι Μάλλον, κυρία Μπιενκόφσκα, ε, κυρίω ε, μεταφέρει τι ευθύνε. Έχουμε εδώ του 2013, έχουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ για το retrofit και αν ε, σκεφτούμε ένα λεωφορείο ε, που κάνει το γύρο της ε, πόλης και εκπέμπει καυσαέρια δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα αυτοκίνητα τα οποία δεν ε, κινούνται όλη την ώρα, ε, αλλά το λεωφορείο κινείται συνεχώς. Εσείς ε, μας μιλήσατε ότι σε επίπεδο ΟΗΕ υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί, κανείς δεν το τήρει. Το θέμα είναι πότε εμείς θα υλοποιήσουμε αυτό ή μάλλον πότε εσείς θα υλοποιήσετε αυτό που είχατε υποσχεθεί το 2013. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καπέσσον τώρα για σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στον Επίτροπο ότι η αναφορά που μας έκανε ήταν πάρα πολύ καλή ε, για τα νομοθετήματα που έχετε φέρει σε πέρας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή δουλειά της Κομισιόν, ιδίως στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, σε ό,τι το περιβάλλον. Και μιλήσατε για την πρώτη που έχει επιτευχθεί. Και είπατε ότι έχετε ξεκινήσει και νέα κεφάλαια. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από όλα αυτά που είπατε. Όπως είπε και ο προλαλής σας όμως, συνάδελφος, αν λείπει κάτι, λείπει μια πιο αποφασιστική δράση για το θέμα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Όλο αναβάλλεται, αναβάλλεται ε, το θέμα αυτό, αλλά χρειάζεται αποφασιστικότητα. Γιατί δεν μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για το παρόν. Πρέπει λοιπόν τώρα να δοθούν απαντήσεις και προς τους πολίτες. Κάτι άλλο. Πολιτικής προσ... Το θέμα πολιτικής προστασίας, μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ξέρετε πρωτοβουλία. Δεν αναφερθήκατε. Ε, μπορεί να βοηθήσει ε, για την καταπολέμηση και της κλιματικής αλλαγής και να δώσει ένα μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρώπη. Εμείς εργαζόμαστε ε, σε ό,τι αφορά αυτό το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και η πρόληψη, η ανάλυση των καταστροφών και αναπεριφέρεια συγκεκριμένα περισσότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για την κλιματική αλλαγή. Και γι' αυτό διερωτώ με μήπως θα χρειαζόταν ένα είδο μηχανισμού, ένα παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή που θα συντονίζει όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη μάχη μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Κάτι ακόμη συγκεκριμένο. Σύντομα θα σας μιλήσουμε ε, για τη Δονιάνα, το φυσικό πάρκο στην Ισπανία ε, που είναι στο Natura 2000 ε, και υπάρχει διαδικασία παραβάση από την Κομισιόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρατυπίες ό,τι αφορά ένα project το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή και σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχετε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, λόγω του ότι πρόκειται για τα δίκτυα Natura 2000. Αυτά είχα να πω. Σύντομα θα λάβετε το σχετικό φάκελο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο ο κύριος εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την ε, δική σας την ε, συνεισφορά στην DG Agri όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος, σε ποια σημεία έχετε επιμείνει. Θα μπορούσατε επίσης να μας πείτε αν συμφωνείτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη και να δούμε επίση αν μπορούμε να έχουμε κάποια οικολογική και τεχνολογική καινοτομία για να αυξηθεί η βιοπικιλότητα, για παράδειγμα, για να καταφέρνουμε να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές, για να προστατεύσουμε τη φύση και το είδωρ αλλά για να καταφέρουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητές μας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Ξέρετε ότι η κυκλική οικονομία έχει άμεση σχέση με τη γεωργία. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα αν προκειμένου. Και μπορούμε επίση να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στην ποιότητα του εδάφου. Πιστεύω ότι ε, αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τον κύκλο ζωής μέσα στο έδαφος, τότε τα ωφέλη θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, συγκράτηση και αποθήκευση του ύδατος ε, στο υπέδαφος, θα καταφέρουμε να αποφύγουμε διαρροή ε, νητροδών καθώς επίσης και άλλων επικίνδυνων ουσιών και θα καταφέρουμε εν τέλει να έχουμε και καλύτερες σοδιές και μια καλύτερη γενικότερα γεωργική παραγωγή. Ποια είναι η δική σας η άποψη λοιπόν, ιδίως όσον αφορά τη διάσταση αυτή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριο Χάουστινγκ, ονομάτων των Πρασίνων. Ναι. Κύριε Επίτροπε, σε σύνοχη τη προηγούμενη ερώτηση για την ε, κοινωνική πολιτική, Γνωρίζετε ποιο είναι ο στόχος μας για τη διατήρησή της βιοπικιλότητας ε, για το 2020. Δεν θα τον πετύχουμε αυτό το στόχο αν δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό στην γεωργική πολιτική γιατί πολλές φορές ακολουθούμε λάθος μέτρα ε, στην κοινωνική πολιτική που ουσιαστικά πλήττουν την βιοπικιλότητα. Είναι βέβαια αρμοδιότητα του Επιτρόπου Χόγκαν, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει στη Γεωργία. Είπε ότι δεν θέλει το γενικολογικό προσανατολισμό ο κύριος Χόγκαν πλέον. Τι θα ακολουθήσει όμως, τι αλλακτική υπάρχει. Τι θα γίνει για το περιβάλλον να λέμε ότι πρέπει να κάνουν πιο πολλά οι αγρότες, παραδείγματος χάρη, για τη βιοπικιλότητα. Δεν ξέρω αν διαβάσετε την ε, έκθεση μάτι για την Νότια Αμερική και την αποψήλωση των δασών και για την καλλιέργεια σόγιας. Ακόμη και για, τη για την Ευρωπαϊκή Γεωργία δραματικά τα νούμερα κατά την άποψή μας. Και σε ό,τι αφορά τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το Μαρκοσούρ, δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε εκτός αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. γιατί δεν ε, κάνει αυτά που πρέπει η Νότια Αμερική. Με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τα Γεωργικά Ζητήματα έχετε επαφή και τι κάνετε από κοινού. Παραδείγματο χάρη και σε ό,τι αφορά τη χρήση των ε, φυτοφαρμάκων. Πώ μπορούμε να τα μειώσουμε. Δεν μιλάμε μόνο για την κλειφοζάτη, η τα νεονικοτιμνοειδη αλλα η χρηση των ε, φυτοφαρμάκων αυξάνεται και πρέπει να τηρήσουν ε, τα σχέδια τα οποία έχουν ε, αναλάβει να εφαρμόσουν για μείωση των ε, ζεζανιοκτώνων τα κράτη-μέλη. Είναι κάποια τα οποία κάνουν κάτι, αλλά άλλα δεν έχουν κάνει τίποτα. Πώς κρίνετε σε όλα αυτά και τι θα κάνετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κύριο Σπεντιτσίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθουμε στο ζήτημα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί και στο παρελθόν, γιατί στη σύνοδο αυτή για την ποιότητα του αέρα στις 30 Ιανουαρίου φάνηκε ότι τα 130 πόλεις από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη παραβιάσει όλες τα ανώτατα όρια τα οποία προβλέπονται. Οι δύο, 7 χώρες έχουν ε, παραβιάσει την, τις, επι, τις, τα νότατα ώρα διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν άλλες πόλεις οι οποίες έχουν παραβιάσει τα νότατα ώρα τα οποία προβλέπονται για άλλα επικίνδυνα αέρια. Ε, καταλαβαίνετε ότι βέβαια θα πρέπει ε, ήδη στα τέλη Απριλίου να εκδικαστούν οι υποθέσει αυτέ από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να μα πείτε συγκεκριμένα ποιε είναι οι χώρε αυτέ και επίση. ε, ποια είναι τα ποσά αυτά τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν από τις πόλεις αυτές. Γιατί αυτή τη στιγμή το τίμημα το πληρώνουν κυρίως οι πολίτες. Έχουμε ένα μηχανισμό που από τη μία πλευρά προσπαθεί να παρακολουθεί τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν ακολουθούν τους κανόνες και επί των οποίων επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις, ωραία αυτό, αλλά από την άλλη πολλές φορές τις κυρώσεις τελικά οι πολίτες τις πληρώνουν με το τίμημα της υγείας τους τελικά. Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας σε παραβάση μια λύση, μια μέθοδος η οποία να είναι πιο δίκαιη για τους πολίτες και να μην ζημιώνει, να μην επιβαρύνει τόσο πολύ τους πολίτες, την η πολιτική είναι αυτή που φταίνε και όχι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Thank you very much. That concludes our... Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο ο πρώτος κύκλος ερωτήσεων. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε κύριε Επίτροπε. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που έθεσε ο Πίτερ. Ο αριθμός για τον οποίο μιλάμε. Συμφωνώ. Τα γεγονότα είναι ε, απαράδεκτα, όχι οι αριθμοί έχουν διευκρινιστεί οι αριθμοί. Προκείται για τον αριθμό πρόωρων θανάτων. Υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ατόμων που πάσουν από χρόνιες ασθένειες. Ναι, θα συνεχίσουμε τις σχετικές δράσεις, όπως σας είπα. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες Μπορώ να απευθυνθώ στα κράτη-μέλη ή όχι, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση αν, η, ε, αν στην πράξη δεν υπάρχει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και σε ό,τι αφορά το retrofitting συμφωνώ μαζί σας. οι διαδικασίες επί παραβάση είναι ίστατη λύση. Στο Παρίσι διοργανώθηκε το φόρουμ για το καθαρό αέρα, έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις, ε, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, τρεις φορές ε, φέτος έχουμε συνεργαστεί και έχουμε ενθαρρύνει τις βέλτιστες ε, πρακτικές. Συνεχίζουμε λοιπόν την υποστήριξη σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Κάπερσον, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα. Ναι, πρέπει να αναλάβουμε δράση και ήδη ξεκινάμε αργά ουσιαστικά γιατί κάποιοι από αυτούς τους στόχους έπρεπε να είχαν επιτευχθεί ήδη από το το 2010. Πράγματι ε, υπάρχει έκτακτη ανάγκη, συμφωνώ. Και σε ό,τι αφορά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, όταν αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, συνήθως μιλάμε ε, για την υποστήριξη των δράσεων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η νομοθεσία μας πρέπει να εφαρμόζεται γιατί η νομοθεσία για το, ε, για το περιβάλλον μπορεί να αποτρέψει τις ε, φυσικές καταστροφές. Και όταν μιλάμε για νομοθεσία για το περιβάλλον, μιλάμε για την αποτροπή ε, φυσικών καταστροφών κυρίως, μεταξύ άλλων που έχουν μεγάλο τίμημα, υψηλό τίμημα και οικονομικό και από ανθρώπινης απόψεως. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τη βιοπικιλότητα. Συγχαίρομαι την Ισπανία γιατί πραγματικά η Ισπανία κινητοποιείται. Τελευταία ε, δράση στην οποία συμμετείχα στην Ισπανία ήταν μια δράση για την κυκλική οικονομία, ε, μια δέσμη μέτρων που υπεγράφει από ε, μεγάλο αριθμό παραγόντων. Και σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, πιστεύω ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα, τρεις μελέτες για την κατάσταση του περιβάλλοντος, η ε, διάμεση αξιολόγηση μεταξύ άλλων, μας λένε ότι έχουμε ξεφύγει από τους στόχους μας και υπάρχει μια γενικότερη τάση. Και η βασική αιτία είναι η γεωργία. Για ποιο λόγο, γιατί η κοινή γεωργική πολιτική και οι πράσινες χρηματοδοτήσεις δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από το Ευρωπαϊκό Ελληνικτικό Συνέδριο. Όταν μιλάμε για την μόλυνση του περιβάλλοντος, του εδάφους, η, ε, τα λοιπάσματα είναι η μεγαλύτερη αιτία μόλυνσης, ρήπανσης των ε, ωκεανών. Αυτή τη στιγμή στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογούμε την κοινή πολιτική, ενδιάμεση αξιολόγηση και και να ορίσουμε τα, ε, τις δράσεις για την επόμενη ευταετία και θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας και σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα και την κοινή γεωργική πολιτική, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τις επικίνδυνες πρακτικές και να χρηματοδοτούμε όσες επιφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την κοινή γεωργική πολιτική η επικοινωνία και σχετικά με την ε, κυκλική οικονομία μεταξύ άλλων και την ασφάλεια τροφίμων ε, συμπεριλαμβάνει πολλές ε, υποσχέσεις για το μέλλον και συμφωνώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και στην καινοτομία πρέπει ε, η κυκλική οικονομία να ενταχθεί σε πολλές ε, δράσεις ε, κυκλικής οικονομίας και να ε, την υποστηρίξει. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του εδάφους, πράγματι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε, η υποβάθμιση, ο κατακαιρματισμός, όπως το είπατε κι εσείς άλλωστε. Ε, νομίζω ότι ο κύριος Χάσλιν και έκανε τα ίδια σχόλια σχετικά με την βιοπικιλότητα, την κοινή γεωργική πολιτική και τα φυτοφάρμακα. Σε ό,τι αφορά τα ε, σχόλια του κυρίου Πιαντιτσίν, τα ίδια έχω να πω. Όταν μιλάμε για την ποιότητα του αέρα, εστιάζουμε κυρίως στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις, αλλά από το 2014 έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επί ε, κατά 13 κρατών μελών. Κατά δύο κρατών ε, η διαδικασία αφορά την ποιότητα του αέρα. Ε, αναφέρθηκα και στον δίκτυ ποιότητας του αέρα. Πρόκειται για πολύ σημαντικό εργαλείο για τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί η ποιότητα του αέρα ε, επιδρά σημαντικά σε ποιότητα ζωής των πολιτών. Με τον ένα ή τον άλλο ε, τρόπο μπορούν οι πολίτες να ε, παρακολουθούν την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε στο, δρομολογήσαμε στο Παρίσι πέρσι στο Clean Air Forum. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχετε ένα λεπτό ο καθένας. Η κυρία Γκροστέτ έχει πρώτα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ανεφερθήκατε στη βιοπικιλότητα στην επαρχία. Έχουμε μια έκθεση του CNRS και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας που αναφέρεται στο ότι εξαφανίζονται πάρα πολύ σημαντικοί πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές εκείνες που καλλιεργούνται στη Γαλλική Ήπεθρο μόνο τότε κάνατε κάποια σχετική αναφορά, πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει κάποιο απολογισμό σε σχέση με την οδηγία για τα ενδιαιτήματα, κυρίω για τα πτηνά, προκειμένου η οδηγία αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική. Επίση, από την άλλη, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη στρατηγική εκείνη την οποία θα δημοσιεύσει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει να κάνει με την επίπτωση φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον μα. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μεταξύ άλλων και στα πλαίσια τη ε, αναθεώρηση των ε, φυτοφαρμάκων και στο, στην επίπτωση που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να καταγράφουμε με έναν τρόπο πιο εναρμονισμένο τον κίνδυνο που α, ενέχουν συγκεκριμένε ουσίε για το περιβάλλον. Καθότι όμω το σύστημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολυπλοκό, θα ήθελα να γνωρίζω αν αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τα φάρμακα αυτά είναι κάτι το οποίο σα έχει απασχολήσει αυτή τη στιγμή και αν επί του ζητήματο αυτού θα δώσετε συγκεκριμένε απαντήσει με τη νέα ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μία ερώτηση όσον αφορά τα δάση. Τα δάση είναι και αυτά οικοσυστήματα πάρα πολύ σημαντικά για το περιβάλλον. Όπω το ξέρετε, ήδη από πέρυσι, εξαιτία των πολύ σημαντικών κλιματικών αλλαγών, αλλά και κυρίω κάποιων ενδημικών προβλημάτων διαχείριση των δασών, τα δάση στην Πορτογαλία και εν γέννη στη Μεσόγειο επλήγησαν πάρα πολύ από σημαντικότατε πυρκαγιέ. Υπάρχει μία η εταιρική σχέση για την προστασία των δασών. Έγινε online μία έρευνα για το ζήτημα αυτό και πάρα πολλοί συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ ενό είδου πορτογαλικού δέντρου που θεωρείται ένα από τα πιο αρχαία δέντρα τα οποία εφίστανται στον πλανήτη μα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε όλο και περισσότερο μια βιώσιμη στρατηγική για τα δάση. Θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δεσμεύσουμε περισσότερα κονδύλια για τα δάση. Μπορούμε επίσης να εκμεταλλευτούμε περισσότερο την ενέργεια την οποία θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε μέσω της βιομάζας. Εγώ είμαι υπέρ της χρησιμοποίησης αυτής της μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα πολύ συγκεκριμένο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει γιατί θα μπορούσε να επιφέρει πολλά θετικά για το περιβάλλον. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση. Μπορούμε εδώ πέρα να συνδυάσουμε λίγο περισσότερο την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα δασικά υπολείμματα τα οποία βρίσκουν μέσα στα δάση. Ο κύριος Λαβή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Εγώ θα μιλήσω για το νερό, για τα ύδατα σε σχέση με τα όσα είπατε εσείς και με τα όσα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Είχαμε ζητήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μια αναθεώρηση των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται και εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ σε μία παράμετρο η οποία χρησιμοποιείται, όπου που βλέπετε ένα μιλίγραμμα ανά λίτρο για τις επικίνδυνες ουσίες που έχουμε στο νερό. 2,4 μιλιγκράμμ είναι αυτή τη στιγμή το ανώτατο όριο το οποίο προβλέπεται. Καταλαβαίνετε ότι ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποδεχθούμε ένα τόσο μια τόσο υψηλή περιεκτικότητα, ιδίως όσον αφορά τα ύδατα αυτά τα οποία βρίσκονται κοντά σε ηφαίστεια. Εγώ αναφέρομαι περισσότερο στη δική μου την περιοχή, στην ε, Σικελία, όπου είχε στηθεί μια εξαίρεση από την παράμετρο αυτή. Θα ήθελα λοιπόν, είχα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μου είχε πει ότι στα πλαίσια τη αναθεώρηση τη σχετική οδηγία θα προβλεπόταν και μία αναθεώρηση των παραμέτρων αυτών και των ανώτων ορίων. Αυτό όμω δεν έγινε στην πράξη. Ακόμα και το ίδιο το κείμενο το οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο πρώτερο ανώτατο όριο, ενώ ο ίδιος, ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτή τη στιγμή έχει προβλέψει διαφορετικά όρια και ουσιαστικά έχει υποβάλει διαφορετικά επιστημονικά δεδομένα. Μήπως θα πρέπει να γίνει μια εναρμόνιση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βόλκαν έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που επηρεάζει βέβαια το έδαφος, καθώς επίσης και τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη από το 2000 στη στρατηγική, ε, μάλλον μέχρι το 2020, θα μπορούμε να έχουμε όλο και περισσότερο εκπομπές διοξιδίου του αζότου από τα πλοία, από τα σκάφη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα μέσα τα οποία έχουμε στη θέση μας για να περιορίσουμε τις διαρροές αυτές. Μολονότι προβλέπεται ήδη ένα σύστημα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν δοθεί τα απαραίτητα κίνητρα. Μήπως θα έπρεπε εδώ πέρα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ομογενοποιημένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους εφοπλιστές, τους κατόχους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις προκειμένου τα σκάφη να γίνουν πιο φιλοπεριβαλλοντικά. Σας είχαμε ζητήσει και στο παρελθόν μέχρι το 2020 να κάνετε κάποιες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Θα θέλω λοιπόν να γνωρίζω αν σχεδιάζετε αυτή τη στιγμή να κάνετε κάτι τέτοιο ιδίως γνωρίζοντας, όπως το βλέπουμε όλοι τελικά ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η μόλυνση της ατμόσφαιρας σε πάρα πολλές πόλεις. Η κυρία Γκαρντίν έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, πολύ σύντομα. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το ΕΛΚΑ όσον αφορά την διαχείριση των μικρών πελαγικών ειδών στην Αδριατική. Σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν και πριν από λίγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια παρουσίασε κάποια δεδομένα βάσει των οποίων θα έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί το πρώτο σχέδιο που υπήρχε για τη μείωση της αλίας στην περιοχή της Εδιαρτικής. Μα υφίστανται, κύριε Επίτροπε, και πολύ διαφορετικοί τρόποι, εναλλακτικοί τρόποι, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να προστατεύσουμε την ε, βιομάζα αυτή των ε, ειδών αυτών που απειλούνται τόσο πολύ μέσω του Eco Survey για παράδειγμα. Είπατε κι εσείς κύριε Επίτροπε ότι ε, ενδεχομένως να μπορούσαν να υπάρχουν νέοι μέθοδοι οι οποίοι θα μας βοηθούσαν τελικά να προστατεύσουμε τα ίδια αυτά, να αλλάξουμε τελικά προσέγγιση όσον αφορά την αλία και στην περιοχή της Ιδρατικής, όπως ακριβώς έχει γίνει και στην Βόρεια Θάλασσα, σε διάφορες σκανδιναβικές χώρες, προκειμένου να μπορούμε τελικά να ρυθμίζουμε τις ποσοστώσεις αλίας με βάση τις την υφιστάμενη βιομάζα των ψαριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε βέβαια ότι από την ελευτική αυτή δραστηριότητα εξαρτώνται και πάρα πολλέ οικογένειε. Οπότε θα πρέπει και αυτή η πτυχή και αυτή η διάσταση να ληφθεί υπόψη. Σα ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Σας Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπή για τις προσπάθειες που κάνετε στον τομέα των επικονιαστών. Και χαίρομαι πολύ που... Με ακούτε? Με ακούτε, ωραία, ναι. Χαίρομαι λοιπόν έλεγα που η Κομισιόν ασχολείται με το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το 2010 πολύ κρίσιμο για τη βιοπικιλότητα τελικά θα ξεκινήσει η διαδικασία σε επιπαραβάση κομισιών για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν στη Μεσόγειο, μιλάω για τα μεσογειακά κράτη, τις απαραίτητες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των πτηνών. Έχουμε απώλεια ε, σε, στους και σε 5.000 ειδών πτηνών. Αυτά απειλούν σοβαρά τη βιοπικιλότητα. Είχα επευθύνει σχετική ερώτηση, αλλά πήρα μια γενικόλογη απάντηση. Άρα ρωτώ συγκεκριμένα, τώρα ξεκίνησαν διαδικασίε παραβάση για χώρες που δεν σέβονται την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν την εφαρμόζουν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Κύριε Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχα σηκώσει το χέρι μου πιο πριν. Μάλλον δεν καταγράψατε το αίτημά μου. Ε, κύριε Επίτροπε, Μιλήσατε για τη βιοπικιλότητα, αλλά δεν μιλήσατε για τα μεγάλα σαρκοφάγα και ιδίως για το λύκο. Μάλλον α, μου φαίνεται ότι υποτιμάτε λίγο το πρόβλημα και οι συνεργάτες σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης κάπως υποτιμούν το πρόβλημα ε, και έχουμε ε, μιλήσει για τη διαχείριση, την ανάγκη διαχείρισης των πληθυσμών των ε, λύκων και στο πλαίσιο της προστασίας της φύσης. Ε, η κατάσταση ποια είναι, η πραγματικότητα ποια είναι. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην Ευρώπη για ένα είδος εύλογου μοντέλου διαχείρισης που δεν έχει όμως βρεθεί αυτό το μοντέλο σε ό,τι αφορά ε, τις κατσίκες, ε, τα πρόβατα και άλλα μικρά ε, ζώα. Πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα για να μπορέσει να εφαρμοστεί και στο μέλλον η πολιτική. Έχουμε την ε, επιστροφή των ε, λύκων. Ε, κάποιοι το θέλουν, κάποιοι δεν το θέλουν. Υπάρχουν περιοχές που υπάρχει ένταση τουρισμού και γεωργικών δραστηριοτήτων και η επιστροφή εκεί των λύκων είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει επαρκείς προσπάθειες να μην το Κυρία Ρίντ. Madam Reid. Ah, good afternoon and thank you for coming. Καλησπέρα και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ τον Νοέμβριο του 2017. Δημοσιεύτηκε από ένα κέντρο στη Γερμανία, ε, κέντρο περιβαλλοντικής μελέτης, ε, που μιλάει ότι 10 ε, ποταμοί οφείλονται για το για το 1% της ρήπασης από τα πλαστικά. Οι τέσσερις είναι στην Κίνα, υπάρχει στην Ινδία, υπάρχει στο Πακιστάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξάγει ανατικλωμένο πλαστικό στην Κίνα εδώ και καιρό. Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας αυτής γερμανικής, σταμάτησαν να παίρνουν ε, Κινέζοι ανακυκλωμένο πλαστικό. Αλλά δεν ξέρω μήπως το πλαστικό που καταλήγει στους ωκεανούς από την Κίνα Μήπως το είχαμε στείλει εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα αρχικά για ανακύκλωση. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίδ. Κυρία Σερπίρικ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την ε, αλία με τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και ο προηγούμενος υφυπουργό και ο νυν υπουργό ε, δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και για το μέλλον, που είναι σημαντικό για το μέλλον της ε, αλληλευτικής πολιτικής που πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Πάντα ήσασταν υπέρ αυτού άλλωστε πολλές οικογένειες ε, που εξαρτώνται από την αλία στις κάτω χώρες αναμένουν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να μας οδηγεί η επιστήμη, όχι τα συναισθήματα. Πριν από λίγους ε, μήνες τα αποτελέσματα που ε, δημοσιεύτηκαν τάσσονταν, συμφωνούσαν με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο οι περισσότεροι ευρωβουλευτές δυστυχώς δεν έδωσαν σημασία μιας και αποφασίστηκε πλήρης απαγόρευση η οποία ε, προκάλεσε αντιδράσεις στις κάτω χώρες οι Ολλανδοί πρωτοστατούσαν σε αυτό το τομέα και τώρα που έχει απαγορευτεί αυτή η πρακτική, η συνεργασία είναι πολύ πιο δύσκολη. Αυτό το θέμα είναι καυτό στις κάτω χώρες και όταν μιλάμε για καινοτομίες πρέπει να διασφαλίσουμε τις καλές σχέσεις. Κάποιος άλλος το λόγο, αν όχι. Εσείς κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την κυρία Γκροστέτ. With regards to... Για τα πτηνά. Ιδίω στην Ήπεθρο. Πράγματι, 55% είναι μείωση από το 90% ε, από το 80 και μετά για αλλαγές ε, στις φυσικές συνθήκες λόγω του ανθρώπου και λόγω της γεωργίας. Πρέπει να σας πω ότι δεν αρκεί η βασική νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωση της διάστασης αυτής ε, και θα πρέπει να υπάρξουν σχετικά μέτρα στην κοινωνική πολιτική γιατί αλλιώς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει εκ των προτέρων. για την υλοποίηση, τα αποτελεσματικότητα που είπε κάποιο. Όταν χρειάζεται να κινηθεί η διαδικασία επί παραβάση ώστε ένα κράτο μέλος ε, να ε, εφαρμόσει την οδηγία, να είστε βέβαιοι ότι αυτό γίνεται. Το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν, το κάνουμε τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η τελευταία περίπτωση ήταν νομίζω κατά της Φινλανδίας, στον προηγούμενο κατάλογο για το Άρλαντ και ένα είδος πτηνού στα νησιά Άρλαντ. Σε ό,τι αφορά τα πτηνά όμως, δεν έχουμε μόνο την οδηγία για τα οικοσυστήματα και τα πτηνά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμαστε και με άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων. Θα μπορούσα να σας παραπέμψω στο έργο μας στο πλαίσιο της ε, ομάδας εργασίας ε, στη Μεσόγειο για την ε, λαθροθυρία και σε άλλες συμβάσεις δραστηριοποιούμεθα. Σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις φαρμακευτικές, είναι κάτι που το συζητούμε. Και είμαστε προβλεπτικοί στη δράση μας. Το έργο μας συνεχίζεται και ελπίζω να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Και να συμπεριλάβουμε τις ε, ενώσεις αυτές που έχουν να κάνουν φάρμακα στις διάφορες άλλες επικίνδυνες ενώσεις. Αυτό που είπατε για τα δάση και τη δασοκομεία εθνική αρμοδιότητα η δασοκομεία. Αλλά δραστηριοποιούμαστε και στον τομέα αυτό. Είχαμε την τελευταία διαδικασία, διαδικασία παραβάση στην Πολωνία πέρυσι. Άρα έχουμε ορθά ανοιχτά τα μάτια μας και παρακολουθούμε την κατάσταση και στον τομέα της διαχείρισης των δασών και αναλαμβάνουμε δράση όποτε χρειαστεί. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βιομάζα, βιοενέργεια. Μπορεί να είναι βιώσιμα, μπορεί να είναι βιώσιμα, αλλά όχι πάντα. Και πράγματι υπάρχει το πρόβλημα ότι εκτάσεις μπορεί να καλλιεργούνται για τη βιομάζα και αυτά τα βιοκάψιμα και όχι για την παραγωγή τροφίμων. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν προωθούμε λοιπόν ε, την παραγωγή αυτή. Gianni, Λαβία Λαβία. Θα το δω, θα το μελετήσω. Αυτό που είπατε. Μου δώσαν τώρα μια απάντηση, αλλά καλύτερα να σας τα πω σε κάποια άλλη στιγμή, να σας δώσω μια γραπτή απάντηση. Καταλαβαίνω τη σημασία που έχει το θέμα για εσάς λόγω της Έτνας που είναι η φεστιακή περιοχή, η φεστιογενής ζώνη και επηρεάζεται. Σε ό,τι αφορά το συνάδελφο Βόλκεν ναι, βεβαίως. Το εξετάζουμε το θέμα αυτό για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν μιλάμε μόνο για τις ε, οδικές μεταφορές ή τις χερσές μεταφορές, αλλά και για την αυσιπλοεία, που είναι ε, σημαντικός ε, παράγοντας ρήπανση. Το έχουμε αντιμετωπίσει και συζητήσει πολλές φορές. Έχω συναντήσει τους εφοπλιστές και τα ε, τομέα των ε, κροαζιερών. Ο κλάδος δεν είναι αντίθετος στη ρύθμιση με νομοθεσία, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα εκπομπών, αλλά αυτό που ενδεχομένως να τους απασχολεί είναι να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μέσω του Διεθνούς, Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Γιατί αν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εντάξει, λέμε πάντοτε ότι πρέπει να ε, έχουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό να μας βάλει σε μειονεκτική θέση. Πάντως ε, εργάζομαι και παρακολουθώ το θέμα πολύ στενά με τη συνάλφο τη Βιολέτα Μπούλτς. Σε ό,τι αφορά το πολιετέ σχέδιο στην Αδριατική για τα πελαγικά. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα πρώτα πολιτή προγράμματα στη Μεσόγειο. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Μεσόγειος. Πάνω από το 90% των προθεμάτων της Μεσογείου υπεραλλιεύονται. Είναι αντικείμενο μάλλον υπεραλίευσης. Δεν έχουμε πετύχει κατά το παρελθόν να διαχειριστούμε με τα εχθή αποθέματα τόσο αποτελεσματικό σε άλλες λεκάνες. Ε, τη γνωρίζω τη Μεσόγειο γιατί έρχομαι, κατάγομαι από τη Μεσόγειο. Δυστυχώς οι αλείς θεωρούν ότι όσο λιγότερη είναι νομοθεσία οι τόσο καλύτερα για την κερδοφορία τους. Δεν ισχύει αυτό όμως. Αν δείτε λεκάνες που συμμορφούνται προς τους κανόνες και τι επιστημονικές ε, συμβουλές, η πρόοδο εκεί είναι μεγαλύτερη. Βιολογική πρόοδος σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, αλλά και οικονομική πρόοδος. Είναι πιο κερδοφόρες οι αληφτικέ δραστηριότητες στη Μεσόγειο, όμως ε, μειώνεται το εχθεαπόθεμα και χάνουν και το εισόδημά του οι αλλοί. Άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη Μεσόγειο. Και γι' αυτό ε, έχουμε αυτό το ίσως το πρώτο πολιτέ σχέδιο για τη Μεσόγειο. Τα μεσογειακά κράτη έλεγαν ε, μην επιβάλλετε κανόνες ε, και νομοθεσία που θα είναι μόνο για εμάς. Γιατί οι βορειοαφρικανικές χώρες δεν θα συμμορφούνται, δεν θα υποχρεώνται να συμμορφωθούν προς αυτά τα μέτρα. Τρία κράτη-μέλη αφορά αυτό το σχέδιο, άρα δεν νομίζω ότι θα αποτύχουμε. Κατά το παρελθόν είχαμε τα λεγόμενα input measures που δεν λειτουργήσαν. Γι' αυτό και τώρα επιλέγουμε output measures για τα συγκεκριμένα αυτά αποθέματα. Είμαστε στην φάση της συναπόφασης και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα για μια ακόμη φορά. Η πολύ απλή απάντηση είναι ναι. Θα κινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση, αν και εφόσον διαπιστώσουμε παράνομη δραστηριότητα για τα πτηνά. Και εμεί συνόρφωση με την οδηγία για τα πτηνά. Το έχω κάνει κατά το παρελθόν. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να το κάνω και στο μέλλον. Για τον κύριο Ντόρφμαν. Για τα σαρκοφάγα. Σαρκοβόρα ζώα. Είχαμε και τους υπουργούς περιβάλλοντος που θέλαν να το συζητήσουν. Αλλά τέλος πάντων, να εστιάσουμε στους λύκους. η αύξηση του πληθυσμού των λύκων δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, δύο, τρία κράτη. Και έχω αναθέσει στις υπηρεσίες μου να δουν το θέμα από την ευρωπαϊκή σκοπιά. Ανησυχώ γιατί μου λένε οι υπουργοί περιβάλλοντος ότι πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε. Ίσως είμαστε θύματα της δικίας μας επιτυχίας, γιατί πέτυχαν αυτά τα σχέδια ανάκτησης του πληθυσμού των λύκων, ξανάρθανε οι λύκοι, επιστρέψαν οι λύκοι, αλλά τώρα έχουμε πρόβλημα στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, με τους λύκους. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ενωσιακό ζήτημα στο άμεσο μέλλον, πιο άμεσο, τις επόμενες μια-δύο εβδομάδες. Έχω τρεις υπουργού που έρχονται για να μου μιλήσουν ειδικά για αυτό το θέμα των λύκων. Σε ό,τι αφορά τα πλαστικά και τα θαλάσσια απορρίμματα στους ωκεανούς. Έτσι τα λέμε, θαλάσσια απορρίμματα. Αλλά ουσιαστικά είναι χερσαία απορρίμματα τα οποία καταλήγουν στον ωκεανό. Το 80% των απορριμμάτων αυτών είναι πλαστικά. Πώς καταλήγουν στους ωκεανούς. Μέσω των ποταμών. Και πράγματι υπάρχουν κάποιες χώρες που προσπαθούν και ελπίζω και να επιτυγχάνουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, να ανακόπτουν την ε, κυκλοφορία των πλαστικών στο ποτάμι. Πριν φτάσει στην ωκεανό, σε την Κίνα, έχουμε καλή συνεργασία με την Κίνα, οφείλω να πω, σε ό,τι αφορά τους ωκεανούς. Και συζητήσαμε το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Με Μάλιστα σκεφτήκαμε μήπως μπορούμε για κάποια θέματα να έχουμε συνεργασία. Και μεταξύ αυτών των θεμάτων είναι τα πλαστικά και τα θαλάσσια απορρίμματα. Αυτό που είπατε τώρα για τα πλακτιστικά που εξάγονται από την Ευρώπη στην Κίνα, κατά πόσον καταλήγουν στους ωκεανούς, δεν το αποκλείω, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει τώρα απαγόρευση εισαγωγών ε, ευρωπαϊκών πλαστικών απορριμμάτων στην Κίνα και αυτό νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να ξεκινήσουν, η Ευρώπη δηλαδή, να ξεκινήσει να ανακυκλώνει τα δικά της απόβητα και απορρίμματα. Λέμε ότι είναι ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα αγαθό τα πλαστικά απορρίμματα. Άρα γιατί να τα στέλνουμε αλλού και να μην τα αξιοποιούμε εδώ. I would like to get resolved. not the... Πρέπει να δούμε επίσης τα τεχνικά μέτρα. Για το ΠΑΛΣ. Που ε, υπερκέρασε όλη τη συζήτηση, επισκέψε όλη τη συζήτηση για τα τεχνικά μέτρα. Τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και ελπίζω να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα στον τριμέρι διάλογο. Υπάρχουν επιστημονικές συμβουλές, πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη μας, έτσι πιστεύω. Αλλιώς δεν θα είμαστε επιτυχείς στη διαχείριση της κοινής ελευτικής πολιτικής. gives us results. If you look at... Το δείχνει η εμπειρία μας. Σε ό,τι αφορά τη μέγιστη ε, βιώσιμη απόδειξη, για παράδειγμα, ε, όταν ακολουθούμε τις επιστημονικές συμβουλές, τα καταφέρνουμε καλά. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γίνεται γιατί ακριβώς ακολουθούμε τις επιστημονικές συμβουλές. Ελπίζω για τα τεχνικά μέτρα να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Σα uh, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για το χρόνο που μας αφιερώσατε, για όλη αυτή τη συζήτηση μπορέσαμε να κάνουμε μαζί σας. Νομίζω ότι και οι συνάδελφοι συμφωνούν ότι είναι πάντα πολύ επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων που έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Προσβλέπουμε λοιπόν στην επόμενη συνάντησή μα Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο, καλή τύχη στη συνέχεια των εργασιών σας. Um, uh, λοιπόν, ας προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Ας κάνουμε κάποιες διοικητικές λοιπόν ανακοινώσεις μέχρι το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη. Στην, την Τετάρτη 27 Μαρτίου από τις 2 το μεσημέρι και μετά θα γίνει με ένα εργαστήριο της Επιτροπής μας για τα πρότυπα εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα από το 2020 και μετά όσον αφορά τα νέα οχήματα και νέα φορτηγά. Μπορείτε όλοι να συμμετέχετε στις 26 Απριλίου το απόγευμα. Ξέρετε ότι είχαμε κλείσει μια αίθουσα προκειμένου να γίνει απογευματινή συνεδρίαση, η οποία όμω δεν θα γίνει. Θα γίνει κανονικά η πρωινή μα συνεδρίαση εκείνη την ημέρα, αλλά είστε ελεύθεροι το απόγευμα. Δεν προβλέπεται απογευματινή συνεδρίαση για τις 26 Απριλίου. Έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες για σήμερα και βέβαια ο φάκελος ε, ε, των εγγράφων είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου η συνεδρίασή μας. Έχουμε πείτε και τις συστάσεις ε, των συντονιστών, σας έχουν διανεμηθεί. Αν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Και βέβαια έχετε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 1ης Φεβρουαρίου και της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου. Πάλι αν μέχρι τα τέλη της συνεδρίασής μας δεν υποβληθούν αντιρρήσεις θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά αυτά. Τώρα, εν συνεχεία, προβλέπεται μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντανιέλ Βιώτη, ο οποίος είναι ο εισηγητής για τον προπολογισμό της Επιτροπής του 2019. Προχωρήσαμε όμως ε, λίγο γρηγορότερα από ό,τι προβλεπόταν, επομένως θα πρέπει να το περιμένουμε λιγάκι ακόμα. Και έπειτα στις 5 ε, έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά το ζήτημα της ε, διπλωματίας για τις κλιματικές αλλαγές. Σας ε, καλώ να παραμείνετε και να συμμετάσχετε και στη συζήτηση αυτή, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Περιμένουμε λοιπόν τον ε, κύριο Βιώτη και φαντάζομαι ότι σε μερικά λεπτά θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μαζί του την ανταλλαγή απόψεων. Well, uh, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, συνταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντανιέλ Βιώτη. Καλώ ήλθατε. Ο κύριος Βιώτη είναι ο συγητής για τον προπολογισμό της Επιτροπής του 2019, τμήμα 3, όπως ενέκριναν και οι συντονιστές, η συμβολή της Επιτροπής μας ΕΝΒΗ για τον, ε, την εντολή που θα δοθεί για τον τρίλογο του Ιουλίου θα γίνει μέσω επιστολής και τον Ιούλιο, 3 Ιουλίου θα συζητήσουμε επίσης και την γνωμοδότηση την οποία θα υποβάλει η Επιτροπή μας, ενώ στις 30 Αυγούστου θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση αυτή. Εγώ υποφαινόμενη είμαι η εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή προς την Επιτροπή Προπολογισμών. Να δώσω πρώτα όμως το λόγο στον κύριο Βιώτη, ή μήπω να πω κάτι εν είδη εισαγωγή Όχι. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο κατευθείαν στον κύριο Βιώτη και στη συνέχεια μπορούμε να υποβάλουμε παρατηρήσεις, να κάνουμε ερωτήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που διεξάγω εγώ όσον αφορά τον προπολογισμό. Επομένω και εγώ έχω να μάθω από εσά, όχι μόνο εσεί από μένα. Θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγα λεπτά, αλλά κυρίω να ακούσω εγώ τα δικά σα αιτήματα, τα αιτήματα τη Επιτροπή Περιβάλλοντο προ την Επιτροπή Προπολογισμών και ακριβώ αυτή την τακτική θα ακολουθήσω και με τι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρω να συγκεντρώσω περισσότερα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι ήδη έχετε δει τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίναμε στην προηγούμενη σύνοδο Ολομελίας του Μαρτίου όσον αφορά δηλαδή το προπολογισμό του 2019, στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές προσπαθήσαμε να δώσουμε πολύ σημαντική έμφαση και στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Λέμε δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αρχίσει να ανησυχεί πάρα πολύ για το ζήτημα το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αποσύρθηκαν από τη Συμφωνία των Παρισίων και ανησυχεί το Κοινοβούλιο για τις ε, ενδεχόμενες επιπτώσεις που αυτό θα έχει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Επίσης, στα πλαίσια των κατευθυντήριων αυτών γραμμών θελήσαμε να θέσουμε κάποιες βασικές προτεραιότητες που έχει προωθήσει και στο παρελθόν και η δική σας η Επιτροπή. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο 20% ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε δηλαδή το 20% του κοινωνικού προπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να δίδεται για, την, για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Και ιδίω να χρησιμοποιήσουμε και τα ποσά εκείνα τα οποία δεν έχουν επενδυθεί στα πλαίσια του εφιστάμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο επεξεργαστήκαμε και βέβαια κάνουμε και αναφορές σε προγράμματα όπως το LIFE, το e-potential, καθώς επίσης και άλλα προγράμματα. Δεδομένου στις εργασίες που έχει γίνει από την Επιτροπή σας και των προτεραιοτήτων που έχετε προβάλει και, σε, και για άλλα προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Λεγγύης για παράδειγμα, και βλέπω και τον αρμόδιο συγκητή τον κύριο Λαβία, ο οποίος ασχολείται και με το ζήτημα της μεταφοράς της EMA στο Άμστερνταμ. Για τα ζητήματα λοιπόν αυτά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να ακούσω τη δική σας την Επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και να συμπεριλάβω κατά αυτόν τον τρόπο τη συνεισφορά σα στην τελική έκθεση που θα γίνει με τον προπολογισμό, πράγμα το οποίο θα γίνει επίσημα και μέσω τη γνωμοδότησή σα. Αύριο θα έχουμε τι πρώτε επαφέ με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τον προπολογισμό 2019 και η βασική μου πρόθεση είναι πέρα από την επίσημη μορφή της συνεργασίας μας, πέρα από την τυπική μάλλον μορφή της συνεργασίας μας, να έχουμε και μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ ημών, όταν θα έχουμε πλέον επισήμως το σχέδιο προπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου τότε θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι προτεραιότητες ανά χορτοφυλάκιο. Το πιο σημαντικό είναι το σχέδιο προπολογισμού του 2019 στο μέτρο του δυνατού να τα αποκρίνεται στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πεπισμένη ότι ζητήματα όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η δημόσια υγεία, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών αποτελούν ανησυχίες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Επομένω, τα νότα όρια που προβλέπονται στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να τηρηθούν απόλυτα και οποιαδήποτε τροποποίηση για να μειωθεί να μειωθούν οι σχετικές γραμμές του προπολογισμού θα πρέπει να απορριφθεί. τα προγράμματα LIFE, καθώς επίσης και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι προγράμματα πολύ σημαντικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραμεριστούν, με συγχωρείτε, για να προωθηθούν άλλα προγράμματα. Επίσης, η απαραίτητη χρηματοδότηση θα πρέπει να δοθεί και για την βιώσιμη προστασία της βιοπικιλότητας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε πιο βιώσιμη χρηματοδότηση προκειμένου να προωθηθεί γενικότερα η βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις ε, τελευταίες εξελίξεις ε, στον τομέα αυτό. Όσον αφορά το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης ε, και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Το ζήτημα αυτό απασχολεί όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καλύτερη δηλαδή διαχείριση των πόρων θα πρέπει να αποτελεί α, ε, οριζόνιο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι μόνο αν έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση θα καταφέρουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να μεταβούμε τελικά προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε, όπως είπατε, το στόχο αυτό, ένα τουλάχιστον 20% του κοινοτικού προπολογισμού να προβλέπεται για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών με χρονικό ορίζοντα το 2020, για τα έτη 2019-2020 δηλαδή, και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ως προς αυτό προσβλέπω στην ακρόαση που θα που θα έχουμε στις 21 Απριλίου με την Επιτροπή Προπολογισμών όσον αφορά το κοινωνικό προπολογισμό και τη Συμφωνία των Παρισίων. Τρίτον, σε σχέση με τους εξωτερικούς οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερα στο ζήτημα των περικοπών στον προπολογισμό, που βλέπουμε ότι επηρεάζει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ του εξωτερικού οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω αυτού που εμπίπτουν στι αρμοδιότητε επιτροπή μα, δεδομένου το ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν όλο και περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητε και αυξάνεται το άχθο εργασία του, αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ε, μια αποτελεσματική προσέγγιση σε σχέση με τους οργανισμούς αυτούς. θα πρέπει να τους δώσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Μα ανησυχεί το γεγονό ότι οι περισσότεροι από τους οργανισμούς αυτούς χρειάστηκε να κάνουν σημαντικές περικοπές στο προσωπικό τους τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από το γεγονό ότι αυξήθηκε το άκτος εργασία τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι κατά περίπτωση θα πρέπει να δούμε τους οργανισμούς αυτούς, θα πρέπει να αξιολογήσουμε δηλαδή τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε εξωτερικού τέτοιου οργανισμού. Τέλος, πρέπει να δούμε και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την αποχώρηση του Μένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους οργανισμούς αυτούς εξωτερικούς και όσον αφορά κυρίως τον, τον ΕΜΑ, τον EMA, και πρέπει να δούμε επίσης τι θα γίνει και με τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Πιστεύω ότι θα πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους και να διατηρήσουμε την υφιστάμενη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Αυτές είναι μερικές από τις ε, ανησυχίες που έχουμε, τις βασικές μας προτεραιότητες που έχετε ήδη εσείς εν μέρει αναφέρει στην αρχική σας αυτή παρέμβαση. Μας είπατε δηλαδή ότι ε, υποστηρίζετε κάποιες από τις απόψεις μας αυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει συμφωνία απόψεων προς αυτό. Να δώσω τώρα το λόγο καταρχά στους ε, σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι όμως δεν είναι παρόντες. Επομένω, ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορείτε να του διαβιβάσετε τα όσα είπαμε. Α πάρουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι το λόγο. Κύριο Λαβία πρώτο. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βιώτη για την εργασία που έχει κάνει και που κάνει. Εγώ ασχολήθηκα με το 2013 και το 2014 με τον προπολογισμό. Ήμουν εισηγητής για το 2013 και ο εισηγητής για το 2014. Γνωρίζω λοιπόν ότι το όλο εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ιδίως θα φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας που καλούμαστε να βρούμε μια συμβαστική λύση και να καταφέρουμε τελικά να συγκεράσουμε όλες τις διαφορετικές προσδοκίες, ανάγκες Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρετε να συγκεράσετε αφενό με τι βασικέ προτεραιότητε που έχουν οι επιτροπέ και όσον αφορά συγκεκριμένα τη δική μα επιτροπή, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο στοιχεία και συμφωνώ εδώ πέρα με την πρόεδρο και η συγκήτριά μα. Όσον αφορά του αποκεντρωμένου οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε ότι κάνουμε συνεχώς περικοπές προπολογισμού των οργανισμών αυτών. Από την άλλη πλευρά δίνουμε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στους οργανισμούς αυτούς. Επομένω, ζητούμε από του οργανισμού αυτού όλο και περισσότερα πράγματα, ενώ από την άλλη του επιβάλλουμε χαμηλότερου προπολογισμού. Καταλαβαίνετε ότι μερικέ φορέ αυτό τελικά καθιστά το έργο του πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με του οργανισμού αυτού καταρχά ένα ακόμα ζήτημα που έχει να κάνει με τους οργανισμούς. Καταλαβαίνετε ότι ορισμένοι από αυτούς εξαιτίας του Brexit θα πρέπει να μετακομίσουν. Εδώ βλέπετε όμως ότι ο προπολογισμό λειτουργεί διαφορετικά. Η συμφωνία για το Brexit, από ό,τι φαίνεται, κινείται περισσότερο τώρα προς μία μεταφορά των ε, πόρων εκείνων ε, στα πλαίσια της συμφωνίας ε, Brexit. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ε, η μεταφορά των κονδυλίων αυτών δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με απόφαση που έχουν πάρει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αλλά έχουν έχει να κάνει με την απόφαση που πήρε το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν εμεί ήδη εκ των προτέρων να πάρουμε κάποιε αποφάσει για το πώ θα γίνουν οι απαραίτητε ανακατανομέ κονδυλίων για να προστατευτούν και αυτοί οι οργανισμοί προτού αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει εκ των προτέρων λοιπόν να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για άλλους οργανισμούς και να γίνουν και οι απαραίτητες διαδικασίες μετακόμισης μετεγκατάστασης κάποιων από τους οργανισμούς αυτούς εξαιτίας του Brexit. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν διευθετηθεί όλο αυτό το κομμάτι εκ των προτέρων, δεν μπορούμε έπειτα να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και την ίδια τη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πότς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντικαθιστώ την κυρία Κάτεμπαχ, η οποία θα ήθελε να τονίσει κάποια ζητήματα που θεωρείται είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή των Προπολογισμών. Θα πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει μία ενσωμάτωση της διάστασης της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων σε όλες τις στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει όλο και περισσότερο η ευρωπαϊκή οικονομία να οδηγηθεί προς μία απαλλαγή από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το πρόγραμμα LIFE, τα πολιτή προγράμματα στο τομέα της υγείας, τα οποία εμπίπτουν βέβαια στην αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής θα πρέπει για το 2019, αν μη τι άλλο, να τηρήσουμε τα κονδύλια για τα προγράμματα αυτά στα πρώτερα επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί ο, ο προπολογισμό μας όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα να συνειδητοποιήσουμε ότι στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού αλλά και στα πλαίσια των εξωτερικών οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται συνεχώ οι αρμοδιότητε. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπεται απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να διατηρηθούν εδώ πέρα προπολογισμοί και θα πρέπει να έχουμε μια εξατομικευμένη κατά περίπτωση εξέταση των αναγκών κάθε εξωτερικού οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον οργανισμό EMA αλλά και στον EFSA. Ο EMA θα πρέπει να μετακομίσει, όπω ξέρετε, από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ. Αλλά και για τον EMA και για τον EFSA θα πρέπει να διατηρηθούν οι προπολογισμοί ώστε να καταφέρουμε τελικά να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε κι εσείς οι ίδια και όπως είπε και ο κύριος ε, Λαβία σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τον αίμα. Αν δεν τους δώσουμε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα, ε, θα επηρεαστεί αρνητικά ποιότητα των πυρογνωμόνων. Χρειαζόμαστε όμως τους καλύτερους εμπειρογνώμονες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο προϋπολογισμός να διατηρηθεί και μάλιστα πρέπει να αυξηθεί. Σε ό,τι αφορά το προπολογισμό για την υγεία, θα ήθελα να εστιάσω σε αυτόν. Λυπάμαι, γιατί κάθε φορά που περικόπτουμε δαπάνες, συνήθως πλήττεται ο οτές της υγείας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πελατικά προγράμματα που πρέπει να υποστηρίξουμε. Για παράδειγμα, για την διασταυρούμενη ε, έρευνα για την ε, τρισομία 21 προκειμένου να αποδειχτεί ο συσχετισμός με άλλες παθήσεις όπως η, ε, το αλσχάιμερ και κάποιες μορφές καρκίνου. Υπάρχουν ε, κάποιοι τομείς που δεν έχουν ε, διερευνηθεί ε, επαρκώς και για το συμφέρον όλων των ασθενών θα ήταν καλό να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα έρευνας και χρειάζονται οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Σημαντικό πολύ επίσης το αίτημα κάποιων επιστημόνων που θέλουν να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τρευματολογίας ή τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένα κύκλο ε, ένας κύκλος ε, εμπειρογνωμών ε, σε αυτό το τομέα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις ε, για να δοθούν απαντήσεις ε, σχετικά με τα, τα θύματα, ε, τους επαγγελματίες υγείας, να υπάρξουν έρευνες σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις που απορρέουν από τέτοια τραγικά γεγονότα όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Υπάρχουν πολλά πιλωτικά προγράμματα που πρέπει να υποστηρίξουμε και που ε, θα καταδείξουν την ε, προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάρ, όχι. Νόμιζα ότι είχατε σηκώσει το χέρι. Η κυρία Γιάρλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω ένα πιο γενικό ερώτημα σχετικά με την πολιτική σας προσέγγιση ως ε, εισηγητής. Διάβασα, ε, ε, παρακολούθησα τους τρεις τελευταίους δημοσιονομικούς κύκλους και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου από την περασμένη χρονιά. Συνήθως η Επιτροπή υποβάλλουν προτάσεις, αλλά εν τέλει δεν καταλήγουμε σε μια ικανοποιητική κατηγοριοποίηση των προτεραιοτήτων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι καινούριο να μας πείτε σχετικά με τη διαδικασία. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα πρέπει ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν θέλει να λάβει το λόγο. Έχουμε εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Αν θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Εξετάσαμε ε, πολύ επιμελώς την πρόταση ψηφίσματος και χαιρόμαστε που ε, περιλαμβάνονται όλες οι ανησυχίες μας, οι περισσότερες. Πράγματι, η Συμφωνία των Παρισίων δημιούργησε μια όθηση ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Λυπούμαστε βέβαια για την απόφαση της, των ΗΠΑ να αποχωρήσουν, αλλά αυτό δεν θα μας σταματήσει εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως η Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα να συνεχίσει τις ε, προσπάθειες και να ε, συνεργάζεται και να ε, ενθαρρύνει τις, τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά έχουν συμπεριληφθεί ε, στις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν μετά τη Συμφωνία των Παρισίων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, δεσμεύτηκαν να, να κάνουν κάποιες δράσεις. Λάβαμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδριού Πράγματι, αναφέρει αυτή η έκθεση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν όλοι οι στόχοι. Απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως η Γενική Διεύθυνση Κλίματος και ε, Προπολογισμό ε, συνεχίζουν να έχουν ως στόχο αυτή τη μείωση κατά 20% των εκπομπών και αυτό θα αποτυπωθεί ε, στο προϋπολογισμό για το 2019, 2020. Στόχος μας είναι τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες και να ε, εφαρμόσουν ε, στην πράξη τις δεσμεύσεις τους. Αυτές τις δεσμεύσεις ε, συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα LIFE εν μέρη και στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κομμάτι του επόμενου ενωσιακού προϋπολογισμού και είναι σημαντικό να πείσουμε τις άλλες γενικές διευθύνσεις να υποστηρίξουν ε, τον επόμενο προϋπολογισμό και να διατηρηθούν ε, τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα. Όσο για τα υπόλοιπα, σας είπα, ε, χαιρόμαστε γιατί συμπεριλαμβάνονται οι ανησυχίε μας ε, στην, ε, στο σχέδιο ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για το live. Λέγομαι Αλεξάνδρα Βάκρου από τη ΓΑΜΑ Περιβάλλον. Εμείς αποδίδουμε ε, μεγάλη σημασία στο live και ιδίω στις συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο. Μαζί με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Κλίμα συνεργαζόμαστε για την εκπόνηση μιας νέας πρότασης για το νέο μέσο. ώστε να συμπεριλάβουμε τις αρτικές προτεραιότητες και των δύο γενικών διευθύνσεων στο μέτρο του δυνατού. Ο στόχος μας είναι η προστασία της βιοπικιλότητας, η κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τα είπε και ο Επίτροπος πριν. Θέλουμε όμως να είμαστε και λίγο περισσότερο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τους αναγκαίους πόρους. Θέλουμε να προωθήσουμε τις ενέργειες και με άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περισσότερη ενεργειακή απόδοση και συνεργασία με άλλους εταίρους για πιο βιώσιμα οικονομικά, πιο βιώσιμη χρηματοδότηση. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που αναφέρατε ήταν ακριβώς η χρηματοδότηση. Με τη νέα χρηματοδότηση θα έχουμε κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις που θέλουμε όμως στο δεθμό του να είναι βιώσιμες. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με άλλους εταίρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταθέσουμε σχετική πρόταση. Λίγο πολύ. Αυτά κάνουμε. Επί του παρόντος. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης που δώσω έμφαση στον ε, όλο και μεγαλύτερο ρόλο που παίζουν ε, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία για τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το κλίμα, το περιβάλλον και την υγεία. Δεν το παραγνωρίζουμε το γεγονός αυτό. Γνωρίζουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ιδίω στρατηγικός εταίρος και για τη περιβάλλον και για τη γαμαδέλτα κλίμα σεβάστηκε απολύτω τα τελευταία χρόνια τι περικοπέ 5%. Αυτό επηρέασε το έργο του, το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τον οργανισμό. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες συνέργειες. Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τον αυξανόμενο ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι οργανισμοί αυτοί. Δεν είναι μόνο οι δύο γενικέ διευθύνσει, αλλά και άλλοι ζητούν τεχνική υποστήριξη στον τομέα του διαστήματος, της έρευνας, της γεωπαρατήρησης με αυτά και με αυτά θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάλφο από τη γάμα δέλτα Σαντέ που θα σας πει βέβαια για τα δικά του θέματα. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Κοντεύουμε τελειώσει το τρέχον δημοσιονομικό. Είμαστε ένα χρόνο πριν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία, τα ποσοστά υλοποίηση είναι σχεδόν 100% και το 2019 περιμένουμε να έχουμε λάβει τα προβλεπόμενα ποσά. Αυτά που προβλέπει δηλαδή το πρόγραμμα τη χρηματοδότηση. ότι αυτά τα πιλωτικά πρόγραμμα τι παραπρασκευαστικής ενέργειε, φυσικά και είμαστε έτοιμοι σε αυτό το χρόνο να εξετάσουμε τι προτάσει του Κοινοβουλίου, να δούμε το κατά πόσο είναι εφικτέ οι προτάσει αυτέ. Και φυσικά στηρίζουμε το αίτημα του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά του αποκεντρωμένου οργανισμού που είναι στο χαρτοφυλάκιο του, ε, δικού, τη δική μα γενική ε, διεύθυνση. ε, βιοκτώνα ΕΚΑΕΜΑ. Κύριε Βιώτη, εσείς τώρα έχετε το λόγο για να σχολιάσετε και να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για την ε, συνεισφορά σας αυτή. Πραγματικά με βοηθά πολύ. Να ευχαριστήσω και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και τους αδέλφους βέβαια από την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σημείωσα τις παρεμβάσεις, τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω βέβαια σε όλες, γιατί ξέρετε ότι η διαδικασία επί του προπολογισμού ξεκινά με αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές και όπως είπε και η συνάδελφος Γκέρλινγκ, εμείς κάναμε πρώτα έναν κατάλογο των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμένουμε να δούμε και ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν φτάσει η πρόταση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε θα καταλάβουμε τελικά πώς διαμορφώνεται ή τι προσανατολισμό παίρνει το σχέδιο προπολογισμού. Σίγουρα υπάρχουν δύο θεμελιώδεις πτυχές επί των οποίων νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όσον αφορά το ζήτημα των ε, αποκεντρωμένων οργανισμών. Ξέρετε ότι ο κύριος Γκάιερ, ο οποίος είναι ο μόνιμος εισηγητής για, τις, ε, για τους οργανισμούς αυτούς, θα ενημερωθεί από μέναν για τα όσα είπατε και εγώ θα ασχοληθώ του χρόνου με το ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως το Συμβούλιο, οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων να συνειδητοποιήσουν ότι από τη μία πλευρά ζητούν όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες, όλο και σημαντικότερο έργο από τους οργανισμούς αυτούς, ενώ παράλληλα, όπως είπαμε, επιβάλλουν περικοπές στο προσωπικό και το προπολογισμό τους. Εγώ λέω ουσιαστικά αυτό είπατε και εσείς, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι ο συνάδελφος ε, Λαβία και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με τον προπολογισμό το γνωρίζουν αυτό ότι αποτελεί πλέον επιβεβαιωμένη τάση στο Συμβούλιο αυτό να ζητάει όλο και περισσότερα πράγματα από τα κράτη-μέλη και από τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη να επιβάλλει περικοπές. Θα έλεγα κατεφημισμό ότι θα είναι ενδιαφέρον το έτος αυτό με όλε αυτές τι συζητήσει που θα γίνουν και για το προπολογισμό του 2019, αλλά ξέρετε ότι παράλληλα θα γίνουν και όλες οι συζητήσει για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αναφέρθηκαν σε αυτό και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν το Συμβούλιο πραγματικά προτίθεται να κάνει επενδύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ολοκληρώνοντας να πω ότι οι προτεραιότητες που από κοινού θα επιλέξουμε για τον προπολογισμό του 2019 θα εξαρτηθούν τελικά και από την στάση που θα κρατήσει το Συμβούλιο. Αν δηλαδή θα θέλει πραγματικά να προωθήσει ένα προπολογισμό ανάκαμψης με βασικές δημοσιονομικές φιλόδοξες προοπτικές και θα εξαρτηθεί επίσης και από τη στάση που θα κρατήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πόσο θαραλέο, πόσο στιβαρή θα είναι η στάση του όσον αφορά τις διεκδικήσεις του. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο Απευθύνομαι και προς την πρόεδρο της Επιτροπής σας, η συγγήτρια για τον προπολογισμό, για την Επιτροπή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας το ζητώ αυτό να γράψετε μια πολύ αυστηρή απαιτητική γνωμοδότηση η οποία θα προσπαθήσει να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες δεσμεύσεις από το Συμβούλιο και εγώ δεσμεύομαι να υποστηρίξω αυτή τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βιώτη και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που πήραν ε, μέρος σε αυτή τη συζήτηση, ως τον παρόντες τουλάχιστον.